Σας παρακαλώ πολύ να καθίσετε. Εγώ σήμερα ε, αναπληρώ τον ε, πρόεδρο Αρτουή. Σήμερα λοιπόν προεδρεύω στη θέση του κύριου Αρτουή, ο οποίος θα έρθει λίγο αργότερα. και θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη. Και προτείνουμε μετά τις ψηφορίες να αλλάξει λιγάκι η σειρά, να πάμε από κάτω προς τα πάνω, πρώτα το 11, μετά το 10 και μετά το 9. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις ε, ψηφοφορίες ε, και μετά όπως σας είπα θα ε, ξεκινήσουμε αντίστροφα. Γιατί το καταλαβαίνετε φαντάζομαι δεν θέλω να συζητήσουμε για την έκθεση Αρτούι αν δεν είναι παρόν και φαντάζομαι ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που τον αφορά ε, θα έχει έρθει ή αν δεν έχει έρθει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αυτό δεν έχει σχέση ε, μόνο με το ότι θέλουμε να είμαστε ευγενεί, αλλά και με το ότι σχετικά με αυτή την έκθεση διεξάγονται ε, πραγματεύσει για αναζήτηση συμβιβασμού. Και θέλω η συγητής να μπορεί να μας παρουσιάσει αυτές τις προτάσεις για συμβιβασμό. Δεν έχουμε άλλες ανακοινώσει του Πρόεδρου, άρα λοιπόν αν συμφωνείτε κι εσείς να περάσουμε είναι ψηφοφορία. Και θα έλεγα να εξετάσουμε πρώτα την έκθεση Όλμπριχ και το ΜΑ Πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφωνία. Ο κύριος Ολμπριχ είπε ότι λείπει, δεν έχει, μάλλον δεν έχει, α, τη βρήκε, τη βρήκε την κάρτα του, πολύ ωραία. Λοιπόν, το πρόβλημα με τον κύριο Αρτουηλή και άρα δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε όταν θα φτάσουμε στην έκθεση του. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Einer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 Λοιπόν, και άλλη δοκιμαστική ψηφοφορία γιατί προέκυψε κάποιο πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στην, ε, στην πραγματική ψηφοφορία. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε τον κατάλογο ψηφοφορίας ε, των ε, σοσιαλιστών που θα βοηθήσει. Δεν ξέρω αν το θέλετε αυτό. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τσεχόφσκι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολύ ωραία. Έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η πέντε του κυρίου Συναδεινού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλφα. α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συγγνώμη, έχει περάσει η ώρα, έκανα και λάθος. Ως εκ τούτου καταπίπτουν οι 6 και οι 11, οι 7 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 9 υπέρ, Νομίζω υπάρχει μία προφορική τροπολογία και θα ήθελα να γνωρίζω ε, κατά πόσον συμφωνεί η συγγήτρια, αλλά δεν είναι παρούσα κυρία Νηριάδο, κύριος Ομαζή, ε, μήπως μπορείτε να μας πείτε ε, κατά πόσον ε, συμφωνεί η ομάδα σας. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε για την τροπολογία χωρίς την προστίκη. Ποιο συμφωνεί με την κυρία Νηριάντα, την 9 παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κύριε Στεχόφσκι, λυπάμαι, υπέρ, η 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ως εκ τούτου καταπίπτουν οι επόμενες από 18 μέχρι 20 και συνεχίζουμε με την 21. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 23 υπέρ. Η 23 καταπίπτει. Η 24... Η 22 καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. Γκρίναμε την 21. Άρα νομίζω ότι έκανα καλά. Η 24 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στην ε, προφορική τροπολογία για την παράγραφο 6. Οι συγκεκριτές προφανώς είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και άλλη προφορική τροπολογία των εισηγητών για την παράγραφο 9 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται η 39 υπέρ εγκρίθηκε η 39 υπέρ κατά Ε, ποιο είναι παρακαλώ κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Θέλετε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 40 παρακαλώ. Υπέρ. Η 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία των εισηγητών για την παράγραφο 15β. Ποιος θέλει παρακαλώ να εγκριθεί. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 50. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται η 51. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η 52. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ως εκ τούτου καταπίπτει 26, 53, 54 και 55 και η τελευταία είναι 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Συγχαρητήρια στους, ε, στην εισηγήτρια, στους εισηγητές μάλλον. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Ε, Νιγκρέσκου είναι ο εισηγητής και περνάμε στην, ε, στη ψηφοφορία τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω μερικοί δεν ψήφισαν καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε η 8 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11 υπέρ, μισό λεπτό, καταπίπτει. Πάμε στην 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Zwei er fehlen noch, einer fehlt noch, jetzt nochmal komplett schließen. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα... Θέλετε, κύριε Αρτουή, να κάνω εγώ την ψηφοφορία για την έκθεσή σας. Αν μπορείτε να μου δώσετε και ένα κατάλογο ψηφοφορίας, παρακαλώ, απευθύνομαι στην πολιτική μου ομάδα.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, το τρένο από το Παρίσι στο Στρασβούργο καθυστέρησε και ευχαριστώ τον κύριο Γκάιερ, ο οποίος ε, με αντικατέστησε στο πρώτο σκέλος των ψηφοφοριών. Δυσκολευτήκαμε λίγο να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμβιβασμό για την ε, έκθεση που μου αναθέσετε για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Με τους συντονιστές και τους κοιόδης ε, εισηγητές ε, καταλήξαμε σε νέες συμβιβαστικέ προτάσεις ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες μας να κάνουν αντίγραφα και να σας τα διανύμουν. Προτείνω, εάν θέλετε, να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία για τις, ε, τον προπολογισμό, τις μεταφορές, ε, αιτήματα μεταφορών. Να δώσω το λόγο στον ε, Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τις διάφορες μεταφορές. Έχουμε την 23, η οποία είναι μια συνολική μεταφορά, την οποία συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ε, υποεκτέλεση και υπάρχει διορθωτικός προϋπολογισμός ε, όπου ε, δίνονται 7,3 δις ευρώ. Σε αυτή την υποαπορρόφηση Έχουμε 855.900.000 που βρήκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν τρόπο να τα επαναδιαθέσει ώστε να μην χαθούν και να χρησιμοποιηθούν. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της ε, συνολικής μεταφοράς και προτείνω να εγκρίνεται. Δεν ξέρω αν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη, στην 24. Αυτή η μεταφορά είναι μια μεταφορά για τη χρηματοδοτική συνεισφορά για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και την Κινητοποίηση. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα και θα ψηφιστεί για την Εστονία. Α, συγγνώμη, ψηφίστηκε, ψηφίστηκε. 1.131.358.000 ευρώ είναι το ποσό. Προτείνεται επίσης 20,3 εκατομμύρια να πάνε στην, στις συνταξιοδοτήσεις, έτσι να καλύψουμε κάποιες επιπλέον ανάγκες για την επικαιροποίηση των ε, συνταξιοδοτήσεων ε, που έγινε τον Ιούλιο του 2015. Προτείνω να εγκρίνουμε και αυτή τη μεταφορά. Το 29 τώρα είναι για την ενίσχυση κατά 10 εκατομμύρια του μέσου για την ειρήνη και τη σταθερότητα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε κάποιες δράσεις οι οποίες είναι εξελίξει αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, στην Τινησία, στην Ιορδανία και ίσως και στην Καμπόν. Το ποσό προέρχεται από το κεφάλαιο εξωτερικής πολιτικής και ε, πολιτική, κοινής ε, πολιτικής και δεν έχει υπάρξει επαρκής απορρόφησης. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε και αυτό το κονδύλι. Μία τελευταία μεταφορά, το 30. Εδώ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουμε και πάλι το μέσο γειτονία 71,5 εκατομμύρια για τους εκτοπισμένους Σύρους πρόσφυγες ε, στις γειτονικές χώρες της Συρίας. Η χρήση προβλέπεται από τη μακροπιστωτική χρηματοδότηση του τομέα της αλίας που δεν έχει απορροφηθεί. Θα υπάρξει κατάλληλη αντιστάθμιση από το Ταμείο Μάντα. Όσον αφορά το θέμα αυτό, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μου πει τι μέτρα ε, λαμβάνει αυτή τη στιγμή προκειμένου να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερα χρήματα στο καταπίστευμα, διότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαθέτει τα κονδύλια, οι δεσμεύσεις των κρατών μελών για τα καταπιστεύματα δεν ε, υλοποιούνται και το ερώτημα είναι πού βρίσκεται η κατάσταση, τι χρήματα διαθέτουν τα κράτη-μέλη, θα δώσουν αυτά τα περισσότερα κονδύλια και τι ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συνεισφορά των κρατών μελών. Θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να σας δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια αυτά. θα χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουμε την δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάσκεψη του Λονδίνου Στόχος είναι η συμβολή στην δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων όσων έχουν πληγεί από την κρίση στη Συρία και στη Συρία και σε γειτονικέ χώρες όπως ο Λίβανος. Με ρωτήσατε τι ακριβώ θα χρηματοδοτηθεί. Πρόκειται για προγράμματα εκπαίδευσης, πρόσβαση στην υγεία, βελτίωση των υποδομών για ε, το πόσιμο νερό, την βελτίωση της αντοχής στην οικονομία, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και την βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της εκπαίδευσης ε, θα είναι η συνεισφορά σημαντική έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο που δέθηκε στη διάσκεψη του Λονδίνου να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ο... Τα χρήματα αυτά θα μεταφερθούν μέσω του τεύματο Μαντάτ. Ε, αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή παρόλο που οι ε, ανέρχονται στα 384 εκατομμύρια, ε, λιγότερο από 80 είναι διαθέσιμα. Επομένω, είναι σημαντική αυτή η έγκριση τη μεταφορά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σύντομα αυτά τα, αυτά τα χρήματα. Το ερώτημά μου όμω είναι, λέει ο Πρόεδρο, εάν τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται στι επιδιώξει τη Επιτροπή, στου στόχου που θέτει η Επιτροπή. Η απάντηση του εισηγητή. Θα ήθελα μια... να μου επιβεβαιώσετε αν τα στοιχεία τα αριθμητικά είναι σωστά. Εάν ε, δεν απατώμε, 69 με 70 εκατομμύρια έχουν δώσει στο Ταμείο Μαντάτ, τα κράτη-μέλη. Ενώ στον προπολογισμό είχαν εγγραφεί 795 εκατομμύρια. Και θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε αν αυτά τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου είναι σωστά και αν ναι, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω μία πρόταση να κάνω. Υπάρχει σχετική παράγραφος στο ψήφισμα για τον προεπολογισμό ε, Αυτά τα κονδύλια ε, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς όπως έχει προβλεφθεί και όπως μπορεί να συμβάλλει αυτή η μεταφορά έτσι ώστε να ε, βοηθηθούν οι γειτονικές χώρες της Συρίας. Όταν όμως θα έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια, τότε προτείνω η Κομισιόν να καλέσει τα κράτη-μέλη να ξαναγεμίσουν αυτό το ταμείο και εμείς μετά θα διπλασιάσουμε. Δηλαδή, ανάλογα με το τι θα καταβάλουν τα κράτη-μέλη, από εκεί θα εξαρτηθεί και το ε, πόσα θα καταβάλουμε εμείς. Εμείς θα καταβάλουμε το 100% αυτού που θα καταβάλουν τα κράτη-μέλη για να διπλασιαστεί ε, το ποσό. Αυτό είναι το αντίθετο ακριβώ από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή κάπου τα κράτη-μέλη ε, να υπόσχονται αυτές οι υποσχέσεις τις ενημερωνόμεθα και της πληροφορούμεθα από τις εφημερίδες. Μετά εμείς ε, καταβάλουμε έγκαιρα ε, τα ποσά που προβλέπεται και τα κράτη-μέλη δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να γεμίσουν αυτό τον κορβανά και εμείς να ε, δεσμευτούμε να διπλασιάσουμε το ποσό. Όπως και να έχει συνάδελφοι, δεν θα το ρυθμίσουμε απόψε. Ε, τίθεται το ζήτημα. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ο Γενικός Εισηγητή για το 2016 για τον προπολογισμό έχει θετική άποψη για τις πέντε προτάσεις μεταφορά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την 23. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ναι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εκρίνεται 33 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. 24. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. τη ψηφοφορίας εγκρίνεται. 30 ψήφοι υπέρ, 8 κατά μια αποχή. 28. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ, 5 κατά μία αποχή. 29 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 34 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 2 αποχέ. Περνάμε τώρα στα υπόλοιπα τμήματα. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν τέσσερα αιτήματα. Πρώτον, ένα αίτημα από την ΕΟΚΕ να μεταφερθούν χρήματα από το κονδύλι για τις, ε, το μισθολογικό προς τις αποζημιώσεις για ε, κάλυψη ενός υπαλλήλου για τον μήνα του Δεκεμβρίου τα επόμενα πέντε χρόνια υπολογίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί να αντιταθούμε σε αυτό. Το επόμενο είναι έτοιμο από το δικαστήριο. Για 55.000 για ε, μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων, ε, τρέχοντα έξοδα αυτά, δεν βλέπω το λόγο να αντιτεθούμε. Τώρα, το επόμενο αίτημα, 870.000 για έξοδα για την βελτίωση της ασφάλειας των κτηρίων και την δημιουργία, μάλλον την, ε, τη μηχανογράφηση και τη βελτίωση της υποδομής για τη μηχανογράφηση στο νέο κτίριο. Μετά, μια μεταφορά 215.000 από, τον, από τη γραμμή 1000 προς την 1654, ε, πάλι στο δικαστήριο είμαστε, είναι για τους ε, παιδικούς σταθμούς. Και επίσης για κάλυψη, ε, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας του δικαστηρίου με το φορέα συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του. Και πάλι θα πρότεινα να εγκρίνουμε το αίτημα. Ο Πρόεδρος, εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ο κ. Ανιώ έχει ζητήσει το λόγο, θα θεωρήσω ότι εγκρίθηκαν. Ο κ. Ανιώ πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ντιπρέ. Μήπω μπορείτε να επιβεβαιώσετε για το πρώτο αίτημα ότι θα καλύψουν ε, το κονδύλιο αυτό πέντε έτη, ενώ ο κανονισμό προβλέπει ότι το μέγιστο χρονικό διάστημα μπορεί να καλύπτεται είναι πέντε χρόνια. Ακριβώ τι προβλέπετε λοιπόν. Απάντηση. Πράγματι δεν μπορούν να ξεβράσουν τα πέντε χρόνια. Αυτό είναι το μέγιστο όριο, αν δεν απατώ. Με μισό λεπτό να δω λίγο τα έγγραφα. Θα σας δώσω τις πληροφορίες που έχω. 18.000 ευρώ και το Δεκέμβριο, μετά 9.000 και για, τους επόμε... για τα επόμενα πέντε χρόνια 10.500. Αυτά τα στοιχεία μου έχουν δώσει. Ερώτηση. Η ερώτηση είναι όμως για πόσους μήνες θα πληρώνεται αυτός ο υπάλληλος που δεν θα κάνει τίποτα. Εδώ πρόκειται για εφαρμογή του παραρτήματος 4 του κανονισμού των υπαλλήλων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προβλέπει ότι ε, εφαρμόζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος, να ρωτήσουμε ε, μήπως μπορούμε να ζητήσουμε από τον εκπρόσωπο του, της ΕΟΚΕ να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αν μπορεί. Δεν είναι εδώ, δεν παρευρίσκεται πρόσωπο της ΕΟΚΕ. Κύριε Νιώ, θέλετε να επανέλθετε, έχετε... Ναι. Απλώς θέλω να δηλώσω ότι αυτό το αίτημα που μας υποβάλλετε μου φαίνεται λιγάκι σαφές. Ε, σύμφωνα με τους κανονισμούς, αυτό αυτό το πρόσωπο θα είχε την δυνατότητα να λάβει χρήματα επί πέντε χρόνια από την ε, στιγμή που συνταξιοδοτητείται και αναρωτιέμαι γιατί καλύπτουμε περισσότερο χρονικό διάστημα. Και δεν, και δεν μου απαντούν και ακριβώ για πόσους μήνες. Είναι λίγο πιο περίπλοκο γιατί το Δεκέμβριο θα λάβει 18.000 ευρώ. Σα το είπα αυτό και από πριν. Μετά, για τρει μήνες θα συνεχίσει να λαμβάνει υποζημίωση ίση με τον βασικό του μισθό. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Δηλαδή 15.000 το μήνα. Μετά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του και τα χρόνια υπηρεσία. η συνταξιοδότηση είναι το 85% του, βασικού μισθού για το οποίο είχε τους τελευταίους τρει μήνες. Αυτό για 4 με 6 μήνε και για τα επόμενα πέντε χρόνια η σύνταξή του θα ανέρχεται στο 60% του βασικού μισθού. Κύριε Σανιό, το μόνο που έχω να πω είναι αυτός ο κύριος ε, έχει κάνει την τύχη του. Απάντηση. Εν πάση περιπτώσει η υπηρεσία δηλώνει ότι είναι προς ε, προ όφελο τη υπηρεσία αυτή η πολιτική, αυτή η επιλογή, επειδή αν είχε παραμείνει στην υπηρεσία θα είχε, κορίσει, ε, κοστίσει πολύ περισσότερο. Ε, ο πρόεδρο ρωτά, υπάρχει ένσταση ή αντίρρηση σε αυτή τη μεταφορά. Όχι, διαπιστώνω. Μήπω υπάρχει κάποια ένσταση υπό τον, για τι άλλε μεταφορέ, Όχι. Επομένω θεωρούνται εγκριθίζε. Βεβαίω θα καταγραφούν στα πρακτικά οι δηλώσει και τα σχόλια που έγιναν. Ε, κύριε Νιώ, ζητάτε το λόγο. Μήπως ε, θα μπορούσα να ζητήσω να γίνει ψηφοφορία επί αυτών των τεσσάρων μεταφορών. Απάντηση του Πρόεδρου, ναι. Ψηφοφορία για το πρώτο αίτημα μεταφοράς. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Le scrutin est clos. 24 υπέρ, 5 κατά. Για τα άλλα τρία αιτήματα δεν θεωρώ ότι υπάρχει... Κύριε Άγνιου, θέλετε να ψηφίσουμε, θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας αν δεν ψηφίσουμε. Εντάξει, εντάξει για τα άλλα τρία έτσι. Γιατί αντιλήφθηνε ότι το ζήτημα είχε τεθεί για το πρώτο αίτημα. Επομένως, έκλεισε το θέμα για τα αιτήματα μεταφοράς και θα επανέλθουμε στη συζήτηση για τον Γενικό Κανονισμό. Σας διανεμήθηκε μια νέα ε, διατύπωση της Γενικής Συμβαστικής Λύσης για τον κανονισμό 25 88, 96, 97, 102, και το, το, το παράρτημα 6, παραγραφή 4, 3, 4 και το οποίο καλύπτει το 1, 4, 5, 6, 7 ο πρόεδρος συνεχίζει να απαριθμεί τους ε, αριθμούς 72, 70 οι οποίοι βρίσκονται και στη, στην κατάλογο ψηφορίας είναι τροπολογία 1, 4, 5, 6, 7 μέχρι 70 βρίσκονται στην, στην, στην, στον κατάλογο ψηφοφορία. Σα διανεμήθηκε λοιπόν η νέα διατύπωση. Κύριε Φερνάνδε, πολύ γρήγορα, ε, νομίζω ότι το 6β, όπως είναι διατυπωμένο, είχαμε πει ότι θα διαγράψουμε το if appropriate. Άρα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι πρέπει να διαγράψουμε και το if appropriate και να ξεκινάει από το the outcome of the consultation shall be put to the plenary vote κλπ. κλπ. Βάσει του άρθρου 314 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαγράψουμε και το if appropriate. Σωστά, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Κατά... Με αυτό λοιπόν ε, σας έχω ενημερώσει για τη συμβιβαστική τροπολογία. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, να ψηφίσουμε την ε, συμβιβαστική πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία για τις τροπολογίες για την τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλετε να ψηφίσουμε μπλοκ. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Να τις ψηφίσουμε 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, πρόκειται για 7 τροπολογίες. 8 μάλλον τροπολογίες. Τις ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, να τις ψηφίσουμε μπλοκ γιατί βλέπω ότι κάποιοι ε, από την 21 μέχρι και την 43 μπορούν να ψηφιστούν unblock. 21 έως 43. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 45 του κυρίου Ταρά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 3 αποσύρεται. Ψηφίζουμε 267 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 70 του κυρίου Γκάιερ υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Le texte εγκρίνεται. 29 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, 2 αποχές. Ο εισηγητής σας ευχαριστεί. Eh Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Και τώρα θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μόλις μας υπέβαλε την ε, νέα της πρόταση για τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Λογικά θα πρέπει να έχουμε κάτι πιο απλό, πιο ευανάγνωστο για τους χρήστες. Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται εν μέρη σε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουμε έναν ενιαίο κανονισμό για τα δημοσιονομικά ζητήματα και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα και υπάρχουν φυσικά και κάποιες τροποποίησεις για τομεακούς κανονισμούς, 15 τον αριθμό, Υπάρχουν κάποιες κοινέ διατάξεις για τα ταμεία επενδύσεων και για τα διαρθρωτικά ταμεία και για τους ε, κανόνες της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα μας επιτρέψει να έχουμε κάποια πιο σαφιστική αν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης που θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους επίσης της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμένου και επίσης εκπροσώπους της Επιτροπής Γεωργίας, Ήτρε, Απασχόλησης Κοινωνικών υποθέσεων ε, περιφερειακής ανάπτυξης, μεταφορών και τουρισμού που είναι εδώ παρούσες μέσω εκπροσώπων για την παρουσίαση και τη συζήτηση αυτών των κανονισμών. Να ε, καλωσορίσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Καλβίνιο, και να της δώσω το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, δίνετε τη δυνατότητα να σας κάνουμε μια παρουσίαση σήμερα για την πρόταση μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού κανονισμού και των άλλων 15 κανονισμών που ανέφερε ο πρόεδρος στην εισαγωγή του. Θα τα πω στα αγγλικά, διότι έχουμε τις διαφάνειες στα αγγλικά και νομίζω ότι θα είναι πιο λογικό. Για άλλη μια φορά λοιπόν να σας πω πόσο σας ευγνωμονώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε από κοινού με την Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για το θέμα αυτό. Ε, αφιερώσαμε πολλή ενέργεια για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε μια καλή πρόταση, μια πρόταση omnibus για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και 15 άλλων νομοθετημάτων και χαίρομαι που κάνω αυτή την παρουσίαση σήμερα διότι θεωρούμε ότι επίγει να υπάρξει πρόοδος στα διάφορα στοιχεία της ε, δημοσιονομικής αρχής όπως βεβαίως είπε και ο Πρόεδρος, εμείς ακόμα δεν έχουμε λάβει μετάφραση, επομένως επισήμως δεν ξεκινάει η διαδικασία, αλλά ε, το Συμβούλιο έχει προοδεύσει ανεπίσημα, έχουν εξετάσει όλο το κείμενο ήδη και επομένως ε, θέλουμε να ακούσουμε και τι ε, προβλήματα αποσχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σήμερα. Η πρώτη διαφάνεια στην παρουσίαση προσπαθεί απλώς να ε, ε, σχολιάσει αυτό που είπε και ο πρόεδρος Αρτουή. Ότι μέσω αυτή τη πρόταση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν ε, περισσότερο τι καταγγελίε και τα προβλήματα τα οποία μας επεσήμαναν είτε η Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο, είτε το Συμβούλιο, είτε τα, οι ενδιαφερόμενοι, είτε τα κράτη-μέλη. Κυρίω θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε την Άνοιξη, προκειμένου να δούμε πώ θα διαμορφώσουμε την πρόταση. Υπήρξαν πολλέ Θετικέ απαντήσει από πλευρά ενδιαφερομένων όσον αφορά την απλούστευση και την ευελιξία. Κάτι βεβαίω που δεν μα εκπλήσει, διότι αυτέ οι δύο άνοιε είναι κάτι το οποίο ε, όλοι επιθυμούν και είναι τα δύο προβλήματα που έχουν εντοπίσει στο παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπήρξαν κάποια ερωτηματικά για ε, ίσονο σημασία ε, ζητήματα, για παράδειγμα κατά αποκοπήν ποσά. Ο ερευνητικό κλάδο αμφισβητήθηκε, αμφισβήτησε αυτά τα ποσά και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε και θεωρούμε όμως ότι γενικότερα υπήρχε υποστήριξη ε, στην ιδέα πλούστευσης των κανόνων. Όσον αφορά ε, τις αλλαγές, μια βασική αλλαγή που θέλαμε να εισαγάγουμε και που ανέφερε και ο κύριος Αρτούη ε, είναι ότι υπάρχει μια πολύ περίπλοκη πυραμίδα νόμων που ρυθμίζουν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού υπολογισμού. Υπάρχουν οι συνθήκε, οι αποφάσει για του ίδιου πόρου, πολιετέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και σχετικό κανονισμό, διοργανική συμφωνία, ε, δημοσιονομικό κανονισμό, κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνε ανακλάδο. Μετά πρέπει να εγκριθούν ε, πράξει κατεξουσιοδότηση, εσωτερικοί κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, ερμηνευτικά σημειώματα κλπ. Χιλιάδες σελίδε εγγράφων και αυτά μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν κάθε περιθώριο ευελιξία που έχουν για να προσθέσουν περαιτέρω απαιτήσει και ανώτατα όρια ε, για ε, τα θέματα αυτά. Επομένω, νομίζω ότι εδώ κάναμε δραστικέ αλλαγέ. Πρέπει να ξεκινήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είπαμε, και αυτό που πρέπει να θέλουμε να κάνουμε είναι να συγχωνεύσουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα νέο εγχειρίδιο. Και ή δυνατόν να μην υπάρχουν ιδιαιτερότητες για κάθε κλάδο και να φροντίσουμε ο δημοσιονομικός κανόνας να είναι ο βασικός ε, κανόνας, το βασικό βιβλίο με τους κανόνες. Δεν τα καταφέραμε στο 100% αλλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο μπορούμε χωρίς να αλλάξουμε την ισορροπία των διαφόρων τομεακών προβλημάτων. Συγχωνεύσαμε λοιπόν τις ε, ε πράξεις κατεξουσιοδότηση με το δημοσιονομικό κανονισμό και προσπαθούμε να δούμε ασυνέπειες και λοιπά που σημαίνει ότι έχουμε 25% μείωση του κειμένου όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες, το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αυτονόητο βεβαίω ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο τη διαδικασία και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι κατευθυντήριε γραμμέ, του κανόνε σε εθνικό επίπεδο κλπ. Δεν είναι μια διαδικασία που τελειώνει στο δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά μέσω αυτού θα περάσουμε στην απλούστευση. Μία αιμονή που έχουμε και είμαι βέβαιη ότι η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα συμφωνεί είναι ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επιδοναμιώσουμε την υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους κανόνες όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε την ορολογία όσον αφορά την φοροαποφυγή κυρίως για τα χρηματοοικονομικά μέσα και έχουμε επεκτείνει και τους κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων σε όλες τις μορφές διαχείρισης. Άρα έχουμε κλείσει όλα τα πιθανά κενά και έχουμε επεκτείνει τους κανόνες ώστε να μην υπάρχει, όπως σας είπα, κανένα κενό ε, και καμία, κανένα παραθυράκι ε, που θα μπορούσε κάποιος να εκμεταλλευτεί η βασική αρχή της πρότασης είναι να απλουστεύσουμε τα πράγματα, κυρίως για αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Θέλουμε να το επιτύχουμε με διάφορα μέσα, το οποίο θα δείτε σε όλο το δημοσιονομικό κανονισμό, επέκταση της χρήσης κατά προκοπήν ποσών για να υπάρχει μικρότερη γραφειοκρατία και λιγότερα σφάλματα. Αυτό το επανάλαβε το ελεκτικό συνέδριο. Θεωρεί ότι είναι μεγάλη πηγή σφαλμάτων το γεγονός ότι είναι πολύ περίπλοκοι κανόνες και τα συστήματα βασίζονται σε ε, πλήρη αποζημίωση των ποσών αντί να χρησιμοποιούνται κατά ποκοπήν ποσά και απλούστερες μορφές και ε, ε, μας προτείνουν όπου υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα ε, για το σύνολο των ποσών και προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε ή να το επεκτείνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης τη χρήση εθελοντική εργασίας που ζητούσε η κοινότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης προτείνουμε να βελτιωθούν οι κανόνες για τη γεωργία για να διευκολύνουμε την ενίσχυση των νέων γεωργών και επίσης θα περάσουμε σε έναν ενιαίο έλεγχο, ένα single audit. Θα επανέλθω σε αυτό εντός ολίγου γιατί είναι βασικό στοιχείο της απλούστευσης. Επίσης προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε ε, κάποιες συνεισφορές απλουστευμένες οι οποίες δεν έχουν σχέση με κόστος, βασίζονται σε αποτελέσματα σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πληρωμή άμα την παραδώσει. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη δικαιούχοι ενισχύσεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Το να προσπαθήσουμε να περάσουμε απευθείας σε πληρωμές ε, με βάση τα παραδοτέα, δηλαδή άτομα τα οποία ε, ε, τα ίσαμε σε συσίτιο. Δεν θα πρέπει να θα μετράμε τον αριθμό και όχι πόσους, πόσα τρόφιμα χρησιμοποιήθηκαν κλπ. Θα τα βασίζουμε στις συνθήκες ή για παράδειγμα τις συνθήκες που ισχύουν εκ των προτέρων. Όπως σας είπα πριν από λίγο, ο στόχος είναι να διευκολύνουμε τη ζωή των δικαιούχων, αλλά επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να μειώσουμε και τα σφάλματα. Το ελεκτικό συνέδριο έχει επισημάνει ότι κάθε φορά που υπάρχουν ε, πληρωμές βάσει ε, των αποτελεσμάτων, βάσει συγκεκριμένων συνθήκων υπάρχουν ε, χαμηλότερα επίπεδα ασφαλμάτων, υπάρχουν η αρχή της, του και δοσκοπικής ε, δράσης που είναι πάρα πολύ σημαντική διότι δίνει κίνητρα σε δικαιούχους ε, να αναζητούν άλλες πηγές χρηματοδότησης ή να προσπαθούν να αναζητήσουν και κάποια άλλα ωφέλη τα οποία μπορεί να προκύψουν από την επένδυση που γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Επομένω, προσπαθούμε να βελτιώσουμε και αυτή την αρχή και έχουμε ε, απλουστεύσει και τον κανόνα των μη σωρευτικών ποσών για άτομα τα οποία λαμβάνουν πολύ μικρά ποσά. Επίση, έχουμε απλουστευμένε διαδικασίε, υπάρχουν λιγότερε εκθέσει για κόστο ε, το οποίο ε, ισχύει στην πραγματικότητα και επίσης ε, ε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση στα αναλυτικά ποσά τα οποία δίνονται στη συνέχεια για αυτά στις πολύ μικρές περιπτώσεις. Επίση, λάβαμε υπόψη μα πολλέ συστάσει του Ελεκτικού συνεδρίου και ελπίζουμε να μπορέσουμε να μειώσουμε το ποσοστό σφαλμάτων έτσι περαιτέρω. Ένα από τα βασικά στοιχεία ε, που προτείνουμε να απλοποιήσουμε έχει σχέση με τους ελέγχους, εκ των υστέρων ελέγχους ε, και διεξοδικότερους ε, ελέγχους. Πολύ συχνά ακούμε αυτή την αρχή του ενιαίου ελέγχου και όλοι υποτίθεται ότι συμφωνούν, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι γίνονται έλεγχοι δύο, τρεις ή και πέντε φορές επιτόπου από τα διάφορα επίπεδα εφαρμογής και ελέγχου. Επομένως, θέλουμε να υποστηρίξουμε πραγματικά τη μετάβαση σε μία ε, διαδικασία ελέγχου, ενισχύοντας ε, την εμπιστοσύνη ουσιαστικά στις διάφορες αξιολογήσεις. Εάν κάποιο θεωρεί ότι είναι ισοδύναμος ο έλεγχο που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε επιπλέον έλεγχο. Μπορούμε να δεχτούμε τον έλεγχο που έγινε στο κατώτερο επίπεδο. Μπορεί να είναι κράτο μέλο, ένα διεθνή οργανισμό, ένα ευρωπαϊκό οργανισμό αυτό που διεξάγει τον έλεγχο. Αυτό πρέπει να τονίσω ότι το υποστηρίζει ε, με κάποια έκπληξη από πλευρά μου πρέπει να πω το ελεγκτικό συνέδριο γιατί δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η αντίδραση του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά στην πραγματικότητα μας υποστήριξαν ιδίω όταν είπαμε ότι θέλουμε να περάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στον έλεγχο των αποτελεσμάτων και όχι του κόστου το οποίο επισήλθε για να σας εξηγήσω αυτή τη μεταφορά. Ξέρω ότι στο πρόεδρο Αρτουή αρέσουν τα διαγράμματα και το να μπορούμε να τους δείξουμε με απλό τρόπο τα πράγματα. Δεν έχουμε λοιπόν ένα απλό διάγραμμα που δείχνει πώς θα περάσουμε από την παρούσα κατάσταση, όπου έχουμε για παράδειγμα μια κυβερνητική οργάνωση που κάνει μια δράση. Υπάρχει εκ των προτέρων αξιολόγηση. Ένα διεθνή οργανισμό υπάρχει, ο οποίο ασχολείται με αυτέ τι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, η Παγκοσμία Τράπεζα για παράδειγμα. Η δράση χρηματοδοτείται και από άλλου διερωτέ και από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, μπορεί να ελεγχθεί μέχρι και πέντε φορέ η ίδια δράση. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό παράδειγμα, ισχύει στην πραγματικότητα, εφαρμόζεται στην πράξη. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα σύστημα όπου θα υπάρχει εμπιστοσύνη στον αρχικό έλεγχο και άπαξ και υπάρχει ένας εκ των, ε, προτέρων έλεγχος που διασφαλίζει ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει, θα περάσουμε σε έναν έλεγχο, ο οποίος θα γίνει επί τόπου, ένας και μόνον, και όπως σας είπα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει, αν ο έλεγχος γίνεται με βάση τα αποτελέσματα και το, την απόδοση μιας συγκεκριμένη δράσης και όχι τον έλεγχο του αναλυτικού κόστους μέχρι και το τελευταίο σέντ. Τώρα, Απλούστευση για τους δικαιούχους, απλούστευση για τη μείωση των αριθμών των ελέγχων και να μην κάνουμε μόνο έναν έλεγχο και να, μια άλλη δράση που προτείνουμε, μια άλλη αλλαγή, είναι να αυξήσουμε τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων μέσων και των τρόπων διαχείρισης. Ε, μία από τις καταγγελίες που λάβαμε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, διαρθρώσουμε τις διάφορες ενισχύσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Να χρησιμοποιήσουμε διαρθρωτικά ταμεία, για παράδειγμα, μαζί με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, ε, όταν υπάρχει έμεση και άμεση διαχείριση, ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκτέλεση που σημαίνει ότι πρέπει να διπλωσιαστούν τα συστήματα ελέγχων. Αυτό είναι και επαχθέ και αυξάνει τον αριθμό των σφαλμάτων. Θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε την κατάσταση στο δυνατόν περισσότερο, να χρησιμοποιεί κάποιο, για παράδειγμα, διαρθρωτικό ταμείο με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, ε, κοινά ε, συστήματα διαχείριση με άμεσα συστήματα διαχείριση, με συνεργασία με άλλου διεθνεί οργανισμού να χρησιμοποιούμε ένα μόνο τρόπο διαχείρισης για την όλη δράση, είτε είναι άμεση είτε έμεση. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να ε, δώσουμε τη δυνατότητα να, εφαρμοστώσουμε, να εφαρμόσουμε ένα σύνολο κανόνων σε μια δράση όταν ε, μετέχουν διάφορα μέσα χρηματοδότησης. Πιο αποτελεσματική χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων όχι μόνο διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλων εργαλείων, αλλά και διευκόλυνση της χρήσης των ίδιων των χρηματοδοτικών μέσων μέσω απλούστερων κανόνων για τις εκθέσεις. Να μην υπάρχει υποχρέωση η ε, ενδιάμεση να υποβάλουν εκθέσεις για τον κάθε δικαιούχο ενός χρηματοδοτικού μέσου. Βεβαίω, αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ ωραία ιδέα να έχουμε πληροφορίε για κάθε έναν από τον δικαιούχο. Αλλά το κόστο που περιλαμβάνει ε, σημαίνει ότι θα υπάρχουν έντυπα 10 σελίδων που θα πρέπει να συμπληρώσει ο καθένα και τελικά οι πληροφορίε που λαμβάνουμε δεν είναι και τόσο ενδιαφέρουσε από τι στατιστικέ πληροφορίε που έχουμε, αν του εξετάσουμε ω σύνολο και δούμε ποια είναι τα βασικά προφίλ τα οποία ε, είναι δικαιούχοι των χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης, θέλουμε να διευκολύνουμε την επανεπένδυση των ε, κερδών που προκύπτουν από τα χρηματοδοτικά μέσα, να περνάνε αυτά και πάλι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ώστε να αυτοχρηματοδοτούνται σε κάποιο βαθμό. Και θέλουμε επίσης να υπάρχουν και ίσοι όροι μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών ε, οργάνων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βεβαίω και είναι ο προνομιούχο εταίρο, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ο μόνο εταίρο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Να περάσω στα τελευταία στοιχεία της πρότασής μας. Πιο ευέλικτη διαχείριση του προπολογισμού. Αυτό προϋποθέτει και κάποια από τα στοιχεία τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην διάμεση αναθεώρηση, την πρόταση που έγινε. Βλέπω εδώ την κυρία Τωμά και νομίζω ότι ήταν και ο κύριος Όλμπριχτ εδώ προηγουμένως. Τέλος πάντων, να υπάρχει ένα, ε, μια δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα 10% για τις εξωτερικές δράσεις ώστε να έχουμε περισσότερη ευελιξία. Ε, μια ταχύτερη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Λιλεγγύης και του Ταμείου ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ διαμαρτύρεται γιατί είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες σε αυτά τα μέσα επέκταση των ευρωπαϊκών καταπιστευμάτων για να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για εξωτερικές δράσεις, αλλά θεωρητικά τουλάχιστον και για εσωτερικέ δράσεις. Δημιουργία ενός αποθεματικού ταμείου για την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωση που θα ε, πρώτα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πάρει ε, ποσά τα οποία αποδεσμεύονται από τις προηγούμενες χρονιές. Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ε, προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την πρόταση για το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και ε, για τα επόμενα τη δημοσιονομικά ε, πλαίσια θα προτείνουμε να υπάρχει ένα ε, κοινό ταμείο τροφοδότησης το γεγονός ότι έχουμε διάφορα στοιχεία, όπως είπε και ο κύριος Αρτουή, ε, ε, μας δυσκολεύει, επομένως θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση και να υπάρχει κοινή διαχείριση για όλα αυτά τα καταπιστεύματα. Απλούστερες και ε, πιο εύκολες διαδικασίες σε διοικητικό επίπεδο. Δεν θα πω πολλά γι' αυτό, γιατί αυτή είναι εσωτερική μας κουζίνα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη δουλειά της διοίκησης. Τα προηγούμενα ήταν να διευκολύνουμε τη ζωή για τους δικαιούχους. Θέλουμε όμως να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα να υπάρχει και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, ώστε να έχουν και αυτοί λόγο για το πού δαπανούνται στις τοπικές κοινότητες τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τέλος, θέλουμε επίσης να ε, επικεντρωθούμε σε αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ε, βασικό στοιχείο για την Αντιπρόεδρο Γεωργίευε και όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε και τη δυνατότητα πληρωμών βάση απόδοσης, αποτελεσμάτων ή ε, προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται και επίσης έναν εξορθολογισμό των εκθέσεων. Να έχουμε λοιπόν κάποιες εκθέσεις οι οποίες θα δίνονται με το σχέδιο προπολογισμού και ένας εκ των υστέρων αριθμός εκθέσεων που θα προκύπτουν στο τέλος την, ε, την ολοκληρωμένη δέσμη εκθέσεων. Νομίζω ότι υπήρχε παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη δέσμη μέτρων ε, και από ό,τι μου είπαν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερος. Καλό είναι να υπάρχει και λίγη λογική στον τρόπο με τον οποίο υποβάλλουμε εκθέσεις. Με δύο λόγια. Συγγνώμη που τα είπα όλα επί γιατί ήθελα να σας πω όλη την πρόταση. Προτείνουμε λοιπόν ένα όμνιμπους, διότι θεωρούμε ότι δεν είναι λογικό να αλλάξουμε κάτι στο δημοσιονομικό κανονισμό, εάν μετά οι τομεακοί κανόνες θα έρχονται σε αντίθεση με αυτό το οποίο προτείνουμε να πλουστεύσουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν υπάρχει μια διαδικασία ενιαίου ελέγχου στον δημοσιονομικό κανονισμό και ο κανονισμός για τις ε, προμήθειες, για παράδειγμα, δεν ε, λάβει υπόψη αυτό το στοιχείο, τότε δεν απλουστεύουμε τίποτα. Αν προτείνουμε ένα κανόνα για την αποφυγή σύγκρουση συμφερόντος και δεν υπάρχει αυτό στους τομεακούς κανόνες, τότε θα υπάρχουν και πάλι ασυνέπειες ε, στο νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε ένα δημοσιονομικό κανονισμό και εξετάζουμε και 15 άλλα στοιχεία της νομοθεσίας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να γελιόμαστε το 85% αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. Μόνο ένα 15% αφορά του τομεακού κανόνε και κυρίω θα κάνουμε αυτά για να ενισχύσουμε τη συνέπεια τη όλη πρόταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια ενιαία διαδικασία διαπραγμάτευσης, σεβόμενοι πλήρω βεβαίω το πώ θέλουν να το διαχειριστούν τα διάφορα θεσμικά όργανα, αλλά εν τέλει θέλουμε να έχουμε ένα συνακτικό σύνολο κανόνων, το οποίο θα μπορούμε να εξηγήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, παρά το γεγονό ότι ε, είναι και περίπλοκοι κανόνες. Δεν θα πρέπει να είναι εύκολο να δαπανούμε δημόσια κονδύλια, αλλά δεν θα θέλουμε να υπάρχουν περιττές ε, επιβαρύνσεις και για τις διοικήσεις αλλά και για τους δικαιούχους. Όπως σας είπα θέλουμε να έχουμε ε, μια συνεπή θέση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεπή θέση και από πλευρά Συμβουλίου. Τι μελιγενέστε ναι, τώρα. Ελπίζουμε να υπάρχει συμφωνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του έτους να έχει υπάρξει πρόοδο και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε η τελική πολιτική συμφωνία για όλη αυτή τη δέσμη μέτρων του Omnibus να γίνει στα μέσα του επόμενου έτους, στη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας, η οποία ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως και ανυπομονεί να αναλάβει την πρόκληση, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες από 1η Ιανουαρίου του 2018. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, όλοι οι συνάδελφοι μου λένε ότι κάθε φορά που προσπαθήσαμε να πλουστέψουμε, αποτύχαμε παταγωδό, γιατί δεν καταφέραμε να τα κάνουμε στο 100%, διότι όταν γίνεται διαπραγμάτευση για το επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε επικεντρωμένοι αλλού και δεν θα ενδιαφέρονται πολύ ε, οι ε, διάφοροι ενδιαφερόμενοι για την απλούστευση των κανόνων. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να αποσυνδέσουμε τη διαπραγμάτευση των κανόνων με, από τη διαπραγμάτευση των ποσών. Θα αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα πριν από το 2020, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Και λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα είπαν οι ενδιαφερόμενοι, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2020 για να αλλάξουμε του κανόνε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να σα τα παρουσιάσω αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Voilà. ευχαριστώ. Ακούσατε και το χειροκρότημα από τους συναδέλφους για να και νομίζω ότι αυτό σας δείχνει πόσο πολύ εκτίμησαν την παρουσίασή σας οι συνάδελφοι της Επιτροπής Προεπολογισμού. Βεβαίως, θα πρέπει να προσέξουμε να μην απογοητευτεί κανείς από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους. 79% μας λένε ότι επιθυμούν την απλοποίηση. 79% και το ερώτημα που θα τεθεί είναι αν η απλοποίηση που προτείνεται και που θα καταφέρουμε τελικά να κάνουμε ήταν επαρκή. Γιατί όλοι έχουμε τέτοια σχετική εμπειρία και τουλάχιστον προσωπικά το έχω ζήσει επί τόπου διαμαρτύρονται οι δικαιοχοι. Μου λένε ότι είναι απαράδεκτα γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σταματώ εδώ. Ποιος ζητάει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως πάντα βέβαια ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα δούμε λιγάκι πιο προσεκτικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτά που μας παρουσιάζετε σε γενικές γραμμές είναι καλά και γέλασα και λίγο με την παρουσίασή σας γιατί ξέρετε τι κάνατε. Δείξατε σε εμά το Κοινοβούλιο τις ε, δικές μας, τα δικά μας τα γραφήματα. Εμείς τα δείξαμε αυτά πριν από έξι χρόνια στην Κομισιόν, ας πούμε την πυραμίδα. Γιατί και μας μας απασχόλησε το θέμα της περιπλοκότητας και όσοι είναι εδώ αρκετά χρόνια θα γνωρίζουν ότι ε, προσπαθήσαμε να πείσουμε την Κομισιόν για αυτά που μας παρουσιάσατε κι εσείς ε, τώρα, δηλαδή να συνδυάσουμε πολλά πράγματα με τους βασικούς κανόνες. Ε, αυτά που μας είπατε είναι ένα παλιό έτοιμο του Κοινοβουλίου να υπάρχει ένα single rule book και, και μόνο γι' αυτό αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε περισσότερο αυτά που παρουσιάσετε. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν το πίστευαν αυτό και άλλοι συνάδελφοι, γιατί αυτό είναι ένας, ένα παλιό αίτημα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πλουστευτούν οι κανόνες, να μην είναι αντιφατικοί, γιατί αυτή τη στιγμή είναι. Και βέβαια ο δημοσιονομικός κανονισμός ισχύει μόνο για το άμεσο management. Ε, βέβαια το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει τα πάντα και προκύπτουν οι σχετικές ε, παρατηρήσεις. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με αυτά που είπατε. Και έχω επίσης διαπιστώσει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει να κατησυχάσω τις άλλες επιτροπές. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ε, είναι ένας πίνακας με ε, τρεις πυλώνες, αυτά που βλέπετε να κρατάω εδώ. Ε, είναι πολύ εκτεταμένος ο δημοσιονομικός κανονισμός γιατί έχει συμπεριλάβει και τους εφαρμοστικούς κανόνες που σημαίνει ότι τελικά εγώ δεν διαπιστώνω να υπάρχουν και τόσο μεγάλες αλλαγές. Βέβαια το κείμενο έχει αλλάξει σημαντικά, γιατί μέχρι τώρα ε, οι εφαρμοστικές διατάξεις έχουν ενταχθεί στο κείμενο και αυτό είναι καλό γιατί αλλιώς ε, ψάχνουν όλοι να βρουν κάτι ε, και από αυτά τα γενικά ε, δεν βρίσκουν άκρη. Τα πράγματα γίνονται περίπλοκα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτά είναι όλα ικανοποιητικά, αξίζουν τον κόπο και θα ήθελα να καλέσω και να καθησυχάσω όλους τους συναδέλφους από τις ειδικέ επιτροπές. Είναι σημαντικό οι ειδικέ επιτροπές ε, να αναλάβουν την ευθύνη για όλα αυτά, όμως υπάρχει σχέση μεταξύ των πραγμάτων ε, και θεωρώ ότι η δική μας ευθύνη είναι κάπου όλα αυτά να στεφτούν από επιτυχία. Γιατί στο Κυριοβούλιο υπάρχουν ε, τάσεις αυτό να αποσυναρμολογηθεί, να αποσταλεί πίσω στην Κομισιόν, να αφαιρεθούν 15 κανονισμοί αυτό όμως πρέπει να το απορρίψουμε ως πρόταση. Εγώ πιστεύω αυτό θα ήταν λάθος. Αν δεν έχουμε τον κανόνα να βλέπουμε, να έχουμε μια συλλογική εικόνα, σφαιρική εικόνα του θέματος, θα έχουμε χάσει μια ευκαιρία κάτι να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να το δούμε όλο αυτό το θέμα, να δούμε τι ακριβώς εννοείται με κάποιες αλλαγές. Η Κομισιόν είναι εξειδικευμένη στο να απλουσεύει τα πράγματα κυρίως για τον εαυτό της. Εμείς ε, είπαμε ότι η απλούσευση πρέπει να προκύπτει για τους αποδέκτες. Και χωρίς να ξέρω το κείμενο, αν ε, δει κανείς όλα αυτά, εκεί που γίνεται λόγος για τον, την κατάργηση των non-profit rules, ε, άρα δηλαδή μια εκδήλωση η οποία έχει λάβει ενίσχυση των 100.000 κόστισε όμως τελικά μόνο 50.000 μπορεί και ο αποδέκτης να κρατήσει τις υπόλοιπες 50.000. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας τριμώξουν στο μέλλον με σκάνδαλα. Ε, εγώ είμαι υπέρ της απλούστευσης, αλλά υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που πρέπει να τα ε, συζητήσουμε εξαντλητικά. Είδα, ας πούμε, ότι έχετε αλλάξει την ονοματολογία, έχετε εισάγει νέους όρους. Πρέπει κανείς να διερωτηθεί τι ακριβώς εννοείται με όλα αυτά. Το βασικό, η βασική πρόκληση για την Επιτροπή είναι οι άλλες επιτροπές να είναι αυτόνομες, αλλά να δεσμεύονται και από αυτό το σφαιρικό έργο. Ούτε και εγώ θέλω να έχουμε 3.000 τροπολογίες ε, για τη γεωργία. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά για να πετύχει πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι και εγώ προτείνω ε, αυτή η Επιτροπή, επειδή έχει το άρθρο 54, ε, να οργανώσει αυτή η Επιτροπή μια νέα μορφή συνεργασίας. Και αυτό που βρήκα εντυπωσιακό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να επιτύχει αυτές τις αλλαγές. Και θα ήταν κρίμα αυτές οι αλλαγές να αποτύχουν λόγω του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία συμπρόεδρε θα έλεγα μάλιστα, γιατί πρόκειται για ε, κοινή ε, επιτροπή και της Επιτροπής Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και μάλιστα ζητήσαμε με βάση το άρθρο 54 να συμμετέχουν και οι πρόεδροι των υπολείπων ε, εμπλεκομένων επιτροπών, βεβαίως με τις αρμοδιότητες που αναλογείς βγουν στην καθεμιά από αυτές. Ο στόχος βέβαια είναι η απλοποίηση. Και θα μπορούσα να ρωτήσω και την Γενική Διευθύντρια μήπως άλλες διατάξεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την απλοποίηση θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από το Omnibus έτσι ώστε να καταφέρουμε να γίνει ψηφοφορές στις 23 Ιουνίου. Κυρία ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη διότι νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε στο δημοσιονομικό κανονισμό όταν εδώ και 7 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία όπως είπατε και εσείς ε, θα τα δούμε επιτόπου με τους δικαιούχους, μας τα ζητούν οι δικαιούχοι και μας τα επισημαίνουν αυτά. Επομένως θα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, πώς θα διαμορφωθεί η πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα βέβαια που οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπω για παράδειγμα στην παρουσίαση το θέμα τη εθελοντικής εργασίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ήταν πάγιο αίτημα όχι μόνο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξη, αλλά και πολλών άλλων ενώσεων. Για παράδειγμα το Youth Forum που ανέκαθεν ε, ζητούσε να συμπεριληφθεί και αυτό στους ε, λογαριασμούς, αν θέλατε, των οργανώσεων. Το single audit ε, το υπενθύμησε και ο πρόεδρος όταν ήμασταν στα ταξίδια στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Πολλοί μας έλεγαν ότι δεν έγιναν πέντε έλεγχοι όπω μα είπατε εσεί στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμένε φορέ φτάναν και του δέκα και ουσιαστικά περνώντα τη μέρα να συμπληρώνουν έτυπα για τον έλεγχο αντί να ασχολούνται με το αντικείμενο των προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι αποτελεί καλή πρόταση η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα και καλό είναι να βασιζόμαστε στα αποτελέσματα και να δούμε αν υπάρχουν αποτελέσματα ε, και όπως για παράδειγμα στην πρόταση ε, για το Ταμείο για τις πιο ευάλωτες ομάδες ε, θεωρώ ότι είναι καλό και το θεωρώ επίσης θετικό στοιχείο και τη δυνατότητα να συνδυάσουμε ή να διευκολύνουμε το συνδυασμό διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων ενισχύσεων για παράδειγμα από τα διαρθρωτικά ταμεία και το σχέδιο Juncker, το ΕΦΣΙ τώρα γιατί είναι αλήθεια ότι σε πολλές από τις περιοχές μας και σε πολλούς δήμους μας λένε ότι είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα. Και ένα θέμα το οποίο προέκυψε και από την προηγούμενη συζήτηση, όλα τα έσοδα τα οποία μπορούμε να έχουμε από τη σωστή διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ. Είναι κάτι το οποίο βλέπω εδώ και στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σχετίζεται και με αυτό που έλεγε ο πρόεδρο, Δηλαδή υπάρχει ένα γαλαξία ο οποίο βρίσκεται πίσω από τον προπολογισμό. Να υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο θα μα επιτρέπει να τα εξετάσουμε από κοινού και να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτά τα κονδύλια και γιατί τα χρησιμοποιούμε. Προφανώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι λεπτομέρειε τη όλη πρόταση, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για μια πρόταση προ τη σωστή κατεύθυνση και εάν καταφέρουμε επιτέλου να απλουστεύσουμε εκεί που λέμε ότι θα απλουστεύσουμε, γιατί μετά θα αρχίσουν να ανακατεύονται οι διάφορες επιτροπές και θα τα περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο, σίγουρα θα έχουμε προοδεύσει αρκετά και έτσι ε, θα είμαστε και έτοιμοι, όπως είπατε και εσείς, για τις διαπραγματεύσεις του 2020, για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να σταθούμε στα ποσά, γιατί τουλάχιστον θα έχουμε λύσει τα θέματα της απλούστευσης. Καλό κουράγιο σε όσους αναλάβουν το θέμα αυτό και θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή Προπολογισμών και φαντάζομαι και ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πρέπει να κάνει τον έλεγχο που πρέπει, αλλά ο έλεγχος δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Ähm, Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, ε, εάν η Κομισιόν κατορθώσει να περάσει τον single audit, ε, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Κυρία Καμπινή, εσείς επισημάνατε ότι είσαστε σε συμφωνία με το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Βεβαίως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να προσπαθούμε να επιτύχουμε απλούστευση και μετά να έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο και να επικρίνει και να λέει ότι δεν ξέρει ακριβώς ε, ποιο σχολείο στο Αφγανιστάν ε, επιδοτήθηκε από ποιο καταπιστευματικό ταμείο και με ποια ευρωπαϊκά κονδύλια. Νομίζω λοιπόν ότι ως, ευρωπαϊκός, ε, ως ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να συνεργαζόμαστε και εδώ θέλω να πω και τη δεύτερη παρατήρησή μου. Ε, οφείλουμε να ε, προσαρμοζόμαστε, να δεχόμαστε και τις συνέπειες. Γιατί πάρα πολλά από αυτά που προτείνατε ε, είναι πιστικά, δεν μπορεί καν να διαφωνήσει κανείς με όλα αυτά. Όταν όμως γράφεται single reporting, αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί ενδεχομένως ε, να ρωτήσει και την τελευταία λεπτομέρεια κάτι που το κάνει με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Άρα δηλαδή το Κοινοβούλιο ε, δεν θα μπορεί να επιχειρηματολογεί πολιτικά. Και τότε θα μπορεί να πει ότι ξέρετε εμείς αλλιώς τα είχαμε φανταστεί ε, και θα είναι σαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην μπορεί να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση και προς τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου να γνωρίζουμε όλοι μας και ποια είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Εκεί που μιλήσατε για τα revenues και repayments, αυτή τη διαφάνεια, ε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που με ανησυχεί σε αυτή τη διαφάνεια ε, ότι θα μπορούν να κατατίθενται εκθέσεις, πολλές εκθέσεις για το ίδιο θέμα και από το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να μην λειτουργεί σωστά το θέμα του κόστους, ε, της μόχλευσης, ε, ε, του εύρους των εργαλείων. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία κριτικής που μπορεί κανείς να ασκήσει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι δογματικός, δεν λέω ότι το καλύτερο από όλα είναι οι επιδοτήσεις. Και ποτέ δεν έπεσα στην παγίδα που μας έχουν στήσει οι Κομισιόν και το Συμβούλιο οι οποίοι λένε ότι ναι θα πάρετε λιγότερα χρήματα αλλά υπάρχουν τα εργαλεία που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε την κατάσταση. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των χρηματοψηφιακών εργαλείων και μπορεί κανείς να παρέμβει με αυτά για να προβεί σε διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο κύριος Μαραγκάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να υποκύψουμε στην θετική πρόκληση της ε, κυρίας Γενικής Διευθύντριας. Ε, Κι εγώ είμαι διατεθειμένος να υποκύψω. Όταν την ακούω, είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου πριν από 15-20 χρόνια στην ε, αυτόνομη περιφέρεια της Βαρκελόνης και σε άλλες ε, τοπικές αυτοδιοικήσεις, να περάσουμε από το σύστημα των εκτονι... Ε, προτέρων ελέγχων στο σύστημα των εκτονιστέρων ελέγχων, που μόλις ακούσαμε. Πολύ ωραία ως κριτήριο. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτή η επιχείρηση, για να μας ασετέ και να υποκύψουμε, ε, εγώ την βλέπω και με θαυμασμό, αλλά υπάρχουν και πολύ περισσότερα στοιχεία. Έχει αλλάξει η ουσία στα κριτήρια διαχείρισης του ευρωπαϊκού προπολογισμού και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε τουλάχιστον αυτό. Αυτοί που ασχολούνται βεβαίως με το θέμα και θα το αναλάβουν θα πρέπει να εργαστούν πολύ περισσότερο ε, να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τη διαδικασία, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, κυρίω η Επιτροπή μα. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί την οργανωτική αυτονομία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες κάθε επιτροπής θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Και βεβαίως αυτό δεν θα πρέπει να υποκατασταθεί αυτό σε καμία περίπτωση, ούτε να μειώσετε το ρόλο μας. Υπάρχει σχετική τροπολογία στην ε, έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και με την εγγύηση αυτής της αυτονομίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το περιεχόμενο, το αναφέρατε κι εσείς νομίζω, νομίζω το, εκτελεστικό, το ελεγκτικό συνέδριο μας το λέει σαφέστατα. Η κόκκινη γραμμή είναι οι ενισχύσεις και η δανειοδότηση. Γίνεται πλέον δόγμα αυτό και επομένω πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Σίγουρα υπάρχουν ενδιαφέρουσες πτυχές, αλλά είναι και πιο ουσιαστική αλλαγή στη διαχείριση του προπολογισμού. Και εδώ νομίζω πρέπει να είμαστε τουλάχιστον πιο προσεκτικοί και να επαγρυπνεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πολιτική απόφαση. Δεν πρόκειται για τεχνική ή χρηματοοικονομική απόφαση. Δεν ε, είναι και δεν πρέπει να είναι. Και όλα όσα εφαρμόζονται σε συνέπεια αυτής ε, της ε, εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα πρέπει να μπορούν να ελέγχονται, να αναθεωρούνται και φυσικά οποιαδήποτε αλλαγή στα κριτήρια διαχείρισης ενέχει κάποιους κινδύνους, όπως ακριβώς ε, το είπε και το ελεγκτικό συνέδριο και μας προειδοποίησε γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό και να ξέρουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Not going to stay long at this either. I think it's late and people are probably getting tired. Δεν θα ακριβωρήσω, γιατί ίσως οι συνάδελφοι σιγά σιγά κουράζονται. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Ορισμένα από αυτά που ακούσαμε σίγουρα θα πρέπει να τα καλωσορίσουμε, όπω για παράδειγμα η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση των διαδικασιών που βοηθούν του νέου αγρότε. Αλλά όπω είπε και η κυρία Κρέσλα, ο διάβαλο κρύβεται στι λεπτομέρειε και θα πρέπει να προσέξουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν ένα-δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε ήδη από τώρα να εξετάσουμε. Να εξετάσουμε για παράδειγμα, ε, τις ε, νέες ή άλλες, άλλους οργανισμούς τους οποίους προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσουμε αρμοτητής ε, ελέγχου και θα ήθελα να μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αυτό θα γίνεται με τρόπο που να σέβεται τις αρχές του ελέγχου της χρήσης δημοσίου χρήματος και καθώς επίσης και να μου εξηγήσει πώς θα υπόκεινται τέτοιου τύπου έλεγχη στον δημοκρατικό έλεγχο που εξασφαλίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ο κύριος Διπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είναι προφανές ότι έκανα μια υψηλής ποιότητας δουλειά και σίγουρα ε, όσον αφορά και την παρουσίαση. Εγώ δεν είμαι ειδικό στο θέμα. Επομένως δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς καθένα από τα μέτρα που μας προτείνεται θα συνεισφέρει στους στόχους. Όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία. Ταυτόχρονα όμως αναρωτιέμαι μήπως μέσω της ε, συζήτησης για την τροποποίηση των κανονισμών δεν περνούν και κάποια άλλα ιδιαίτερα θέματα. Για παράδειγμα, μια φράση η οποία μου. Μου έκανε εντύπωση authorization of trust funds, η εξουσιοδότηση για την ε, δημιουργία τέτοιων κατασπιστευματικών ταμείων και εγώ θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η σχέση τέτοιων ταμείων με τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Επομένως, στις προτάσεις που μας παρουσιάσατε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την απλοποίηση. Για παράδειγμα, αναφέρεστε στην ε, μεγαλύτερη ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών, citizens engagement, ε, στην ε, μεγαλύτερη συμμετοχή λοιπόν των Ευρωπαίων πολιτών στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. μάλιστα, αλλά αυτό τι σχέση έχει με την απλοποίηση και πώ ακριβώς επίσης σκέφτεστε να το πετύχετε. Κάτι ακόμα για το οποίο θα ήθελα να μου δώσετε διευκρινήσεις. Το πρώτο θέμα ήταν, όπως σας είπα, τα trust fund. Το δεύτερο θέμα για το οποίο θα ήθελα διευκρινήσεις είναι αυτή η έννοια του, που αναφέρεται στο Omnibus για τη μεταφορά χρημάτων από του ενός, ε, από ένα ταμείο σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν είναι σαφέ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι συγκεκριμένο θα σημαίνει, διαφορετικά θα το έχετε συμπεριλάβει. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε ακριβώ λοιπόν τι σημαίνει. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος κι εγώ. Βεβαίως χρειάζεται μια απλοποίηση των διαδικασιών για τις πληρωμές. Το ίδιο πρέπει να ε, συμβεί και με τους, ε, τις διαδικασίες ελέγχου. Και οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να είναι απλοποιημένες. Και αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης στο, στα, ταμεία, στα ταμεία Όμω ορισμένε φορέ πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε μια ε, μεγαλύτερη, σε περισσότερο βάθο ανάλυση για να καταλάβουμε από πού προκύπτουν οι καθυστερήσει. Συχνά δηλαδή διαπιστώνεται μια καθυστέρηση, αλλά δεν γίνεται η ανάλυση ε, που θα μας επέτρεπε να καταλάβουμε τι είναι η προκάλεση. Ο πρόεδρος ζητά κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Με την άδειά σας. Δεν θέλω να πω κι εγώ ορισμένα λόγια. Είμαι ιδιαίτερος ε, θετικά διακείμενο προς την προσπάθεια που κάνετε και χάρηκα με την παρουσίαση και με αυτά που άκουσα αυτήν. Μέσα από δύο-τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα ήθελα να σκεφτούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η απλοποίηση, τι, ακριβώ ακριβώς θα συμβεί αυτή η απλοποίηση. Και θα σας δώσω λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Προσωπικά είχα την εμπειρία ενός πιλωτικού προγράμματος, μικρού πιλωτικού προγράμματος, το οποίο ως πιλωτικό είχε στόχο να πειραματιστεί, να πειραματιστούμε με νέες μεθόδους. Και αντί να επιτρέψουμε αυτόν τον πειραματισμό, ε, βάζουμε τους ε, προτείνοντες, τους δικαιούχους στη μέγενη και τους δυσκολεύουμε σε οποιαδήποτε τους κίνηση. Ε, δεν είναι λογικό όταν γίνεται ένας προ, προ, ε, ε χρησιμοποιείται κάτι καινούριο, γίνεται ένας πειραματισμός, δεν είναι λογικό ότι θα υπάρξουν δυσκολίες. Όταν βλέπουν τις διαδικασίες λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι, απλώς απογοητεύονται και δεν στέλνουν ούτε καν πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσει αυτή, αυτά τα προβλήματα, αυτή η κολυσιεργία στον τομέα των πιλωτικών προγραμμάτων. Μετά, αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι κανόνες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι το αποτέλεσμα προηγουμένων πολιτικών διαπραγματεύσεων και ψηφοφοριών, αλλά μην ξεχνάμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 εμείς θα είμαστε οι υπεύθυνοι. Επομένω, θα πρέπει σύντομα να κινητοποιηθούμε. Γι' αυτό σα ζητώ να μας δώσετε ε, κάποια, συγκεκριμένα παραδείγματα για να είναι ξεκάθαρο και στα μέλη του Κοινοβουλίου αλλά και στους ενδιαφερόμενους, ε, στους δικαιούχου, πώς θα λειτουργήσει η απλοποίηση που προτείνεται. Τώρα βέβαια υπάρχουν και δυσκολίες οι οποίες ε, οφείλονται στην ε, εθνική νομοθεσία. Άλλε δυσκολίε οφείλονται στην εθνική νομοθεσία και άλλε οφείλονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρη διάκριση. Για να μπορούμε να χωρίσουμε την Ιρά το στάρι. Επομένως, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας. Τη βρίσκω εξαιρετική, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε στο τέλος να έχει αποτέλεσμα και να μην είναι απλώς κάτι που κάναμε για τα μάτια του κόσμου. Παρακαλώ, έχετε λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας που έκαναν πολύ κέρδιες παρατηρήσεις πριν απαντήσω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα πρώτα να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για κάτι που κάνουμε για τα μάτια του κόσμου. Πραγματικά έχω γίνει τσιμπούρι στους συναδέλφους μου. Κάθε εβδομάδα τους ρωτάω σε αυτή τη διαδικασία απλοποίησης κάνατε πραγματικά ό,τι μπορούσατε να κάνετε. Και μετά από εμένα έρχεται και η αντιπρόεδρο, η κυρία Γεωργίαβα, η οποία επίση ρωτάει, κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σα. Έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η απλοποίηση ήδη από τα νέα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή που θα ξεκινήσουν να ε, υλοποιούνται έτσι ώστε να λάβουμε και περισσότερες προτάσεις για αυτά. Προσπαθούμε να αυξήσουμε ε, τη, τις δυνατότητες που δίνουμε στους πιθανούς δικαιούχους, χωρίς φυσικά να ε, προτείνουμε ή να επιβάλλουμε μια πλήρη αλλαγή, πλήρη αναθεώρηση του συστήματος. Τώρα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα που ε, τέθησαν για το ζήτημα του μη χαρακτήρα. Η κυρία Κρέσλα έχει δίκιο. Δεν πρέπει να πληρώνουμε περισσότερα από ό,τι έχουν εγκριθεί για ε, μια επιδότηση, για μια ενίσχυση. Από την άλλη υπάρχουν κανόνες που δείχνουν ότι ένας ερευνητή στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να πληρωθεί για ένα άρθρο ε, και δεν έχει κανένα κίνητρο να οργανώσει ε, κάποιο συνέδριο. Γιατί αν το κάνει αυτό θα προκύψει κάποιο κέρδο. Άρα δηλαδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρείται το ανωτοτόριο, δεν θα καταβάλουμε μεγάλα ποσά. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να σκοτώνουμε εκείνα τα προγράμματα που θα είναι επιτυχημένα. Ε, άρα δηλαδή πρέπει κάπως να προσπαθούμε να βρούμε την σωστή ισορροπία για να μην εξαφανίζουμε τα κίνητρα. Άλλοι ε, αναφέρθηκαν στο θέμα της, ε, του reporting, της λογοδοσίας με την ευρύτερη έννοια, αν το καταργήσουμε αυτό, ε, δεν θα υπάρχει κανένα δημοκρατικό έλεγχο. Θέλω να πω ότι εμεί δεν μειώνουμε τον αριθμό των εκθέσεων, απλά εξορθολογίζουμε εκείνου που υπάρχουν στο δημοσιονομικό κανονισμό. Επίση, προσπαθούμε να αποφύγουμε τι επικαλύψει και τελικά αν έχουν ήδη προκύψει κάποιες εκθέσεις, κάποιες αναφορές δεν ε, θα πρέπει ε, να προσθέτουμε κάτι που είναι άχρηστο εκ των υστέρων. Δεν χρειάζεται να παναφευρίσκουμε οτιδήποτε. Και τρίτον, έχουμε ε, καταργήσει την υποχρέωση αναφοράς μεμονωμένων αποδεκτών, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν καταργούμε τη διαφάνεια, του αντίον την ενισχύουμε, τουλάχιστον σε ένα τομέα που είναι τα καταπιστευματικά ταμεία. Σε αυτά λοιπόν προτείνουμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου ε, και το έχω ακούσει επανειλημμένα αυτό σε αυτήν την Επιτροπή. Γιατί έχουμε προτείνει να επεκταθεί αυτή η δυνατότητα και με μια εσωτερική διάσταση, διότι διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι εργαλείο το οποίο πρέπει να προκύψει για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον ίσως ε, να μην υπάρχει αυτό πλέον στο μέλλον και για κάποιες ενέργειες μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση Πάντως όχι γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας κανονικός τρόπος ε, χειρισμού του ευρωπαϊκού ε, προπολισμού. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Πάντως εμείς προτείνουμε να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία. Και υπάρχει μια ερώτηση για το κατά πόσον θα πρέπει να πάμε στο εκ από το εκ των υστέρων στο εκ των προτέρων. Εγώ δεν συμφωνώ ε, αλλάξαμε τους κανόνες με βάση αυτά που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια. Είχαν, υπήρχαν πάρα πολλά έγγραφα που έλεγαν τι θα έπρεπε να μεταφραστεί ε, και μετά εκ των υστέρων έλεγχος και ποσοστό σφάλματος. Εμείς πιστεύουμε ότι αν κάνουμε έλεγχο εκ των προτέρων και ε, θεωρούμε ότι κάποιοι οργανισμοί έχουν παρεμφερείς κανόνες, τότε ε, θα πρέπει ε, να υπάρχει μεγαλύτερη αναλογικότητα. Κατά τα άλλα, Υπήρξε και μία ερώτηση ε, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους εταίρους. Εμείς έχουμε κατά νου τις εθνικές ε, αναπτυξιακές τράπεζες που υπάρχουν σε αρκετά κράτη-μέλη και ε, όπου οι κανόνες είναι παρεμφενείς θα πρέπει αυτοί να είναι ίσως εταίροι μας όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με τον τρόπο που έχουμε συντάξει αυτό το εργαλείο επιθυμούμε να είναι οι οργανισμοί δημόσιοι. Αυτό είχαμε κατά νου όταν συντάξαμε αυτές τις ε, νομοθετικές διατάξεις. Επίσης υπευλήθη μια ερώτηση από τον κύριο Ντεπρέ και θα σας απαντήσω. Εδώ τι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση μιας δέσμευσης την οποία τελικά αποδεικνύεται ένα κράτος μέλος ότι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για να αξιοποιηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Λοιπόν, θα μπορούσε ε, ε, ένα κράτος μέλος να ζητήσει αυτό το χρηματο... Ε, τα χρήματα που υπήρχαν στο χρηματοδοτικό εργαλείο να μεταφερθούν σε ένα άλλο ταμείο κοινοτικό, έτσι ώστε να μην χαθούν τα χρήματα. Όμως δεν, δεν αλλάζει ο τρόπο διαχείριση. Δεν είναι ότι κάτι το οποίο βρισκόταν στην επιμερισμένη διαχείριση το πηγαίνουμε στην άμεση, απλώ προσπαθούμε να διευκολύνουμε το κράτο μέλο. Ναι, μέλος. Δεν είναι ο στόχος μας να αποσύρουμε χρήματα από το χρηματοδοτικό μέσο, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε όταν αυτό είναι, βοηθάει ε, και είναι το σωστό ένα κράτος μέλος. Επίσης, όσον αφορά τη διπλή υποβολή εκθέσεων. Εδώ θέλουμε να την αποφύγουμε, γιατί για παράδειγμα έχω επιστρώσει ότι υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει για τα διαρθρωτικά ταμεία και για τα, ε, τα κοινοτικά ταμεία. Και ε, όταν τι εξετάσουμε σε βάθος, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αλληλεπικαλύψει. για παράδειγμα σε ζητήματα περιβαλλοντικά κτλ και να δεν χρειάζεται να υπάρχουν δύο εκθέσεις για, τα για το ίδιο θέμα μόνο και μόνο επειδή υπήρξε μια μεταφορά χρημάτων από, ένα, ε, από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό σε, σε, σε, ένα ταμείο του κράτους μέλους για παράδειγμα. Τώρα, Ευχαρίστω, όπω πρότεινε ο πρόεδρο τη Επιτροπή σα, να έρθουν εκπρόσωποι ε, τη Επιτροπή για να σα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η απλοποίηση θα λειτουργήσει σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πεδίο. Ε, έχουμε οργανώσει τέτοιου τύπου σεμινάρια για του δικαιούχου και του ενδιαφερόμενου και ευχαρίστω να έρθουμε και εδώ. Και τέλος να σας ε, διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να υπονομεύσουμε την θεσμική αυτονομία και θεσμική ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος παρεμβαίνει. Μήπως θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και εκπροσώπους των τοπικών αρχών σε αυτό το σεμινάριο που αναφέρεται, για να μας πούνε και τη δικιά τους προσέγγιση και τη ε, δικιά τους ε, οπτική γωνία για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η απλοποίηση. Απάντηση. Ναι, ναι, ναι βεβαίως. Έχουμε άμεση ε, επικοινωνία με την Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί Πράγματι, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές, όλους εκείνους που υλοποιούν προγράμματα, ε, ε, χωρίς να ε, διακινδυνεύσουμε βεβαίως τη χρηστή διαχείριση. επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα λοιπόν, δεν έχουμε κανένα στόχο να υπονομεύσουμε τη θεσμική αυτονομία του Κοινοβουλίου, να προσπαθήσουμε να το επηρεάσουμε αλλά θα σας ζητήσω, ε, εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη fast track στα γαλλικά, να έχουμε μια ταχεία διαδικασία, ένα fast track σε αυτή τη συζήτηση για να μην καθυστερήσουμε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και εμείς. Δεν είχαμε καθόλου την υποψία ότι θα προσπαθούσατε να χειραγωγήσετε τη συζήτηση. Υπόσχεται πολλά λοιπόν αυτή η συζήτηση και σίγουρα θα την συνεχίσουμε. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Η κυρία Καλβίνιο θα μας ενημερώσει και πάλι για ε, το, την επιστολή 10. Ε, καλό βράδυ κυρία Γκράσλε. Από 10 Νοεμβρίου επισήμως θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία του τριλόγου. Ε, τροποποιητική επιστολή ε, 1. Είναι το σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη. Έχετε το λόγο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη γιατί είναι πολύ αργά και όπως είπατε δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επιστολή. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο συνήθως ε, υπάρχει μια τροποποιητική επιστολή που είναι η βασική τροποποίηση στην πρόταση του σχεδίου προπολογισμού που έχουμε υποβάλει και συνήθως ο στόχος αυτής της τροποποιητικής επιστολής είναι να περιλαμβάνει τις ε, πιο πρόσφατες ε, πληροφορίες που έχουμε για την εκτέλεση του γεωργικού προπολογισμού. Επειδή ολοκληρώθηκε μόλις η ετήσια εκτέλεση του προπολογισμού και λαμβάνουμε υπόψη και τις δαπάνες, επικαιροποιούμε τον προπολογισμό για την επόμενη χρονιά χρονιά. Φέτος η τροποποιητική επιστολή διαφέρει κατά τη, διότι έχουμε συμπεριλάβει όλες τις προτάσεις που αφορούν το 2017 για να μεταφράσουμε την πρόταση της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης που έχουμε υποβάλει. Υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο τμήμα της επιστολής ε, που αφορά την επικαιροποίηση της ε, δαπάνης για τον ε, γεωργικό τομέα. Αυτό, όπως θα δείτε, είναι κυρίως τα μέτρα τα οποία αναφέρθηκαν για το γαλακτοκομικό τομέα, 500 εκατομμύρια. Επίση, θα θυμάστε ήδη ότι στο σχέδιο προπολογισμού είχαμε συμπεριλέβει 100 εκατομμύρια για τα φρούτα και το προκυπευτικά, αλλά εδώ λαμβάνουμε υπόψη και τα γαλακτοκομικά και τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί και επίσης μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα επιπλέον μέτρα μέσω αυξημένων εσόδων. Επομένω, δεν αλλάζει τίποτα στι δεσμεύσει του σχεδίου προπολογισμού και νομίζω ότι υπήρχε και μείωση των πληρωμών κατά 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθο. Επομένω, όσον αφορά τα συνολικά ποσά, δεν είναι πολύ σημαντική η αλλαγή στο σχέδιο προπολογισμού. Υπάρχουν όμω αυτά τα επιπλέον μέτρα για το γαλακτοκομικό τομέα. Πέραν αυτών, έχουμε συμπεριλάβει και έχουμε ε, στο σχέδιο προπολογισμού και κάποια μέσα για να αυξήσουμε τις δαπάνες, τα λεγόμενα top-up ε, της ε, ε, μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης σε δύο τομείς. Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και μετανάστευση. Όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, προτείνουμε αύξηση κατά 50 εκατομμύρια των δεσμεύσεων υποχρεώσεων για τον ορίζοντα 2020 το κόσμο και το safe transport. Και δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα τώρα για αυτές τις τρεις προτάσεις και τα τρία προγράμματα, διότι ξέρουμε ότι ο κύριος Φερνάνδες ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτά τα προγράμματα και η Επιτροπή Προϋπολογισμών εν και θέλετε να τα ενισχύσετε. Επίσης, θέλετε να ε, πρικοδοτήσετε και την πρόταση για τη σύνδεση ασύρματου διαδικτύου που θα προκύψει από το σύστημα, πρόγραμμα Telecom και 50 εκατομμύρια επιπλέον για το Erasmus Sin, κυρίως στον τομέα της μαθητείας. Ένα πρόγραμμα το οποίο γνωρίζω ότι το υποστηρίζετε πολύ εδώ στην Επιτροπή. Επιπλέον, δεν έχουμε συμπεριλάβει τα το μόνο για το 2017, αλλά δεδομένου και του ε, προγραμματισμού έχουμε λάβει υπόψη μας τα προγράμματα και για το 2020. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ε, επίσης ε, και το συνολικό περιθώριο για τις δεσμεύσεις χρεώσουν. Υπάρχει διαθέσιμο ένα κονδύλιο ακόμα εκεί και προτείνουμε αύξηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση της νεολαίας με επιπλέον ένα δις και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στις δεσμεύσεις υποχρεώσεων στο συνολικό περιθώριο, προτείνουμε μια ε, συμφωνία με το Συμβούλιο ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αυτή την αύξηση του χρόνου όταν θα υπάρχει επιπλέον περιθώριο, θα υπάρχει πρικοδότηση και επομένως θα κάνουμε τις προσαρμογές στην άνοιξη του 2017. Προτείνουμε λοιπόν αμέσω ε, σχέδιο τροποποιητικού προπολογισμού για να συμπεριλάβουμε αυτά τα κονδύλια ε, στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ο δεύτερος μεγάλος κλάδος δράσης είναι η μετανάστευση. Εδώ προτείνουμε 750 εκατομμύρια για την ε, στήριξη της πρότασης πλαίσιο με τις χώρες εταίρους. Ε, υπήρχε μεγάλη υποστήριξη για αυτή τη συνολική στρατηγική την προηγούμενη εβδομάδα που συζητήθηκε πρέπει να πω και αυτό ε, περιλαμβάνει τα 500 εκατομμύρια για το μέσο ανάπτυξης και συνεργασίας, 250 ε, εκατομμύρια για το μέσο κοινωνία. Προτείνουμε επίσης 250 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αυτή τη στιγμή είναι υπό διαπραγμάτευση, και θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση με ε, κάποιες μεταφορές ποσίων ώστε να φτάσουμε στα 375 εκατομμύρια. Και προκειμένου να τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά, προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί και το αποθεματικό ε, για το 2017. Προτείνουμε να ενεργοποιηθούν αυτά τα ποσά από το, αποθεματικό, το περιθώριο του αποθεματικού. Ξέρετε ότι πρέπει να το καθορίσουμε αυτό και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην επιβαρύνουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Προτείνουμε λοιπόν να ξεκινήσουν τα ποσά για το 2017 μέχρι το 2019 με βάση τον τίτλο 2 το 2017 και τον τίτλο 5 το 2018 και 2019. Στην ε, διορθωτική επιστολή προτείνουμε να ενισχύσουμε και τη Europol με 20 επιπλέον θέσεις εργασίας, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις θέσεις οι οποίες προτάθηκαν με το προσχέδιο προπολογισμού του 2017 και να δώσουμε τη δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ακτοφυλακής και Συνοριοφυριακή και την ΕΑΣΟ, την Υπηρεσία Σύλλου, να εκπληρώσουν πλήρως τα καθήκοντά τους και την ανάγκη να προσλάβουν έμπειρο προσωπικό. Επομένως, ε, προτείνονται κάποιες επιπλέον θέσεις εργασίας με βάση το προσχέδιο προπολογισμού και επομένως ο προπολογισμός για τις θέσεις αυτές είναι υψηλότερος. Ε, προτείνουμε επίσης και τρεις αλλαγές όσον αφορά τις διοικητικέ δαπάνες. Πρώτον, να απλουστεύσουμε και να εξορθολογήσουμε ε, διοικητικά, οικονομικά στοιχήματα και συστήματα επιμελητία. Προτείνουμε λοιπόν τα καθήκοντα των τριών ειδικών εκπροσώπων με διπλή ιδιότητα από τον τίτλο 2 στον τίτλο 5. Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον διότι αυτό ήταν προπόθεση από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού τη ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μείωση κατά 15% τον, ε, τον αριθμό του ε, ε, προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Επομένως, μειώνεται η υποχρέωση να υπάρχουν παράλληλες θέσεις εργασίας για διοικητικά καθήκοντα σε αυτές τις συγκεκριμένες αντιπροσωπίες. Δεύτερον, προτείνουμε να το συμπεριλάβουμε στον προπολογισμό και τις υποχρεώσεις ε, για ε, τη μισθοδοσία, δηλαδή να υπάρχει η αρχή της ε, διαδικασίας που περιλαμβάνει τον πληθωρισμό στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και την εξέλιξη της μισθοδοσίας σε 11 κράτη-μέλη. Δεν έχουμε ακόμα τα τελευταία στοιχεία τα οποία αφορούν αυτή την αύξηση των μισθών, αλλά προτείνεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υψηλότερα τα ποσά από αυτά που είχαμε προβλέψει στο προσχέδιο προπολογισμού. Και ε, τέλος, στον τομέα της διοίκησης προτείνουμε να ευθυγραμμίσουμε τον αριθμό θέσεων εργασίας στα σχέδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δύο ε, επιτροπών ε, με βάση τη συμφωνία που επετεύθη στο θέμα αυτό μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Βασικά θεωρούμε ότι αυτή η διορθωτική επιστολή μεταφράζει τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση στην ε, ε, ενδιάμεση διαδικασία προπολογισμού και δεδομένου ότι όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν για τον προπολογισμό του 2016 και το προσχέδιο προπολογισμού για το 2017 και τη διορθωτική επιστολή θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τους δύο βραχίονες της αρχής προπολογισμού και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση για τη διορθωτική επιστολή, η οποία μας δίνει την ε, δυνατότητα τώρα να συζητήσουμε ε, το Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, πάρα πολλά από αυτά που αναφέρονται στη διορθωτική μου επιστολή ε, δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς ε, να τα επικρίνει όταν πρόκειται για την πολιτική, για τη γεωργική πολιτική και για όλα αυτά που έχει ήδη εγγράψει το Κοινοβούλιο ως βούλησή του στο σχέδιο του προϋπολογισμού. προβλέπεται η ενίσχυση των κονδυλίων, το περιμέναμε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι ε, ακολουθήσετε ένα αρκετά επικίνδυνο δρόμο με την έννοια ότι αυτά τα οποία συνδέονται με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο τα εγγράψατε, το Συμβούλιο όμως είναι λιγότερο ευέλικτο από ότι είμαστε εμείς και τελικά ε, θα μπορούσε το Συμβούλιο να περιπλέξει περισσότερο την όλη διαδικασία διότι θα μπορούσε να δεχτεί μόνο τα ε, διοικητικά εργαλεία αλλά ε, να μην προβεί σε ενίσχυση των κονδυλίων. Θέλω αύριο να το ρωτήσω αυτό στην Ολομέλεια, αλλά πρέπει να σα πω ότι ήδη γνωρίζω ποια θα είναι η απάντηση. Όσον αφορά τα ε, εργαλεία ενίσχυσης, ε, χαιρόμαστε για το ότι σε πάρα πολλά σημεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα τις επιφυλάξεις μας σε σχέση με την επαναφορά των προσεγγίσεων πριν από το ΕΦΣΥ Connecting Europe Facility και Horizon 2020, αυτά να τα προβάλλετε περισσότερο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αρκετά ε, ενισχύονται. Εμείς θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν αναφερόταν ότι παίρνουμε αυτά τα χρήματα που υπάρχουν επιπρόσθετα έτσι ώστε να επανέλθουμε στην κατάσταση πρώτου εύση. Κατά τα άλλα, η διαδικασία που προτείνεται είναι ενδιαφέρουσα και όσον αφορά ε, στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, διερωτώθηκα ε, πώς ακριβώς ε, πρέπει κανείς να ερμηνεύσει τα στοιχεία, τους αριθμούς που παρατίθενται. Κατάλαβα ότι το 2017 να το στο μότο δυνατόν το 1 δις. Ε, θα θέλαμε κάτι περισσότερο βέβαια. Αυτό όμως μπορούμε να το διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο κατά πόσον δηλαδή ε, θα πρέπει να ακολουθηθεί η δική μας η κατεύθυνση. Και βασικά ε, στην δημοσιονομική διαδικασία αποφασίσαμε για μια πολιτική βούληση με το Συμβούλιο και ε, ίσως αν αποδειχθεί ότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την ενίσχυση αυτών των ε, κοντιλίων ε, θα πρέπει να συζητήσουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το ποσό. Αυτό που δεν μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτά που προτείνεται στο Global Europe, γιατί είναι λιγάκι μονομερή. στον τριμερή διάλογο τα έθιξα λιγάκι, η ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί επιθυμούμε διακαώς τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν να ενισχυθούν και ε, το μέτρο της ε, έκτακτης βοήθειας να μην είναι το μόνο το οποίο θα μπορεί να ισχύει. Και αυτό ισχύει και για το εργαλείο σταθερότητα και ε, ειρήνη και πολιτική γειτονίας. Εκεί πρέπει να σας πω, οι προτάσεις σας μου φαίνονται αρκετά μονομερείς. Και όταν πρόκειται πολλές από αυτές τις προτάσεις να τις αντικαταστήσετε με ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για Βιώσιμη Ανάπτυξη, φτάνουμε σε αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Εγώ ανησυχώ γιατί αυτό το ταμείο θα μπορούσε να συνδυάσει δύο δυναμίες, δηλαδή την έλλειψη προσθετικότητας την οποία επικρίνουμε ε, στο ΕΨΗ και άλλα εργαλεία τα οποία ενδείκνυνται να επιτύχει κανείς αναπτυξιακά προγράμματα με ενισχύσεις. Θα πρέπει να συζητήσω με τον εισηγητή για το κατά πόσο όλα αυτά μπορούμε να τα στηρίξουμε. je Σας ευχαριστώ. Δυστυχώ συνάδελφο Ταρού, Ταγού πολύ θα ήθελε να ήταν μαζί μα. Απόψε που συζητούμε το θέμα του τρι, τριμερού διαλόγου που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Δυστυχώ αυτό δεν είναι στάθη δυνατό γιατί είχε καθυστέρηση το ε, αεροπλάνο του. Τώρα η ο κύριος Φερνάντες, ο συζητητής για τον προπολογισμό 2017, μήπως έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Μια επιθυμία θα ήθελα να εκφράσω. Εγώ ελπίζω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είναι σύντομα σε θέση να εκφράσει την θέση του, να λάβει θέση επί της διορθωτικής επιστολής η οποία συνδέεται άμεσα με τον προϋπολογισμό 2017. Την οποία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη βεβαίω, αλλά συνδέεται επίσης και με την αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά τα τρία θέματα η διορθωτική επιστολή, ο προπολογισμό 2017 και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και αναθεώρησή του συνδέονται. Γι' αυτό θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα να είναι σε θέση να ξεκινήσει την ε, συζήτηση επί τη ουσία. Ο Πρόεδρο. Και επί αυτού του σημείου θα έλεγα ότι μάλλον δεν μα καθησύχασε η παρουσία του Συμβουλίου στον τριμερή διάλογο. Γιατί είναι άλλε συνθέσει του Συμβουλίου σε καθέναν από τους ε, τριμερεί διαλόγους. Για την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού ε, πλαισίου είναι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ενώ για τον προπολογισμό 2017 είναι το ΕΚΟΦΗΝ. Και όσον αφορά τη διαδικασία, μας είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα μετά την συμφωνία επί του 2017 ε, θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού. Δεν βλέπω κάποιο άλλο να ζητάει το λόγο. Άρα θα θεωρήσω ότι οι ομιλητέ ήταν πολύ ξεκάθαροι στην παρουσίασή τους και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξη, δηλαδή την έκθεση του Χωσέ Εμμανουέλ Φερνάντε. για την πιθανό, πιθανή αναστολή των κυρώσεων που θα μπορούσαν να, να επιβληθούν στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα πει ότι ε, θέλετε να τα κάνω γρήγορα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα τα πω γρήγορα. πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβάλλει κανείς κυρώσεις σε έναν ολόκληρο λαό για να ε, τιμωρήσει μια κυβέρνηση. Η επιβολή μιας ανα, αναστολής ε, ε της ε, χρηματοδότησης από ένα ολόκληρο χρηματοδοτικό ταμείο θα ήταν πολύ σοβαρή. και ευελπιστώ ότι αυτή θα είναι η θέση την οποία ομόφωνα θα υιοθετήσει και η Επιτροπή Προπολογισμού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή και παρά το γεγονό ότι είναι αργά, θα ρωτήσω όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής εάν θεωρούν ότι συμφωνούν με την άποψη του κ. Φερνάντες εάν μπορούμε να δώσουμε την ομόφωνη στήριξή μας σε αυτό που είπε ο κ. Φερνάντες μόλις τώρα. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται ναι. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν και την ε, ημερησία μας διάταξη. 9 και 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες θα είναι η επόμενη μας ε, συνεδρίαση και αν υπό τα διάφορα δεν θέλει κανένα μέλος το λόγο θα θεωρήσω ο αυτή μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ που καθίσατε μέχρι τόσο αργά το βράδυ. Καλή νύχτα.